Και τώρα περνάμε στην κανονική μας εργασία σύμφωνα με την ημερησία διάταξη και πρέπει να πω ότι από πλευράς συντεπαλέστρης εθίγει ένα θέμα υπήρξε ένα αίτημα το οποίο και του κυρίου Σπένσκι και του κυρίου Βάντιμ Τούντορ ζήτησαν να μπορέσουν να επωφεληθούν από το καθεστώς των ε, κοινοβουλευτικών ασυλίων και θα απευθυνθούν τα αιτήματά του στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Τούτων λεχθέντων διαδικαστικό εσείς παρακαλώ. 847 παρακαλώ. Δεν κατάφερα να κατανοήσω με ακούτε. Δεν κατάφερα να καταλάβω αυτά που είπατε. Ο κύριος Magistris ζήτησε, αν κατάλαβα καλά, να μην αρθεί η ασυλία του. Τι είπατε. Κοιτάξτε, ο κύριος Ντεματζίστρης ε, στην χώρα μου είναι ο πρωταθλητής εναντίον της διατήρησης της ε, ασυλίας. Οπότε ίσως να υπάρχει εδώ ένα λάθος στη μεταφορά του νοήματος. Παρακαλώ να διευκρινίσετε αυτό το οποίο είπατε για τον κύριο Ντεματζίστρης. Yes, and that's what you said. It was probably just a problem with the translation. What, what, what It's said? requested to defend his parliamentary immunity under the provisions of the law. Yeah, it was uh, uh, such a, it was such a request. Ένα τέτοιο αίτημα διαβιβάστηκε όπως ανέφερα και πρόκειται να αποφασιστεί, θα αποφασίσει η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου όσοι ήθιστε άρθρο 6 εδάφιο 3 του κανονισμού μας. Ζητήθηκε να <clears throat> προστατευτεί αυτή η ασυλία, όπως θα σας είναι γνωστό. Uh, και περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια, στο, στην ημερήσια διάταξη. Και σύμφωνα με, τον, με το άρθρο 4, εδάφιο 1 και εδάφιο 4, σημειώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή την κατάσταση πραγμάτων και με βάση το άρθρο 3 εδάφιο 2 η κυρία Μόνικα Κλέφερ Πρέντεγκάστ και Σάντο